στη Ζιμπάγκου αγαπητοί συνάδελφοι έχει λήξει και μπορούμε να ψηφίσουμε. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη ψηφοφορία για τον Ai Weiwei. Έχουμε έξι προτάσεις ψηφισμάτων. Τροπολογία 2. Καταρχήν με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Ψηφίσατε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3, πάλι με ονομαστική. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίθηκε. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος. Υπέρ, κατά. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, δεν ψηφίζουμε με ονομαστική. Εγκρίθηκε το ψήφισμα. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο θέμα. Εξόριστη κυβέρνηση και εδώ υπάρχουν έξι προτάσεις. Ξεκινάμε με την πρόταση του EFD. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Το κοινό ψήφισμα. Καταρχήν όμως πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται α, να ελέγξουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά αρχή της ψηφοφορίας ψηφίσατε τέλος της ψηφοφορίας απορρίφθηκε με δύο ψήφους διαφορά τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψηφίζουμε ψηφίσατε τέλος εγκρίθηκε αυτή η τροπολογία ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Τέλος, το τελευταίο θέμα για το οποίο πρέπει να ψηφίσουμε είναι 7 διαφορετικά ψηφίσματα για την Ζιμπάμπουε. Ξεκινάμε με το ψήφισμα της ομάδας EFD. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα έχουμε το κοινό ψήφισμα, παράγραφος 10, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται το αιτιολογική σχέση λάμδα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τελική ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος και εδώ ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Τέλος των ψηφοφοριών, τέλος της συνεδρίασης. Θα σας διαβάσω τώρα μία δήλωση στα τσεχικά. Τα πρακτικά